Ladies Κυρίες και κύριοι σας, καλώς ορίζω. Και πάλι έχουμε αργήσει και πρέπει να προσπαθήσουμε κάποια στιγμή να αρχίζουμε στην ώρα μας. Θα χρειαστεί λίγος χρόνος μέχρι να συνηθίσουν όλοι, αλλά μετά θα τελειώνουμε και στην ώρα μας για να μην τιμωρούμε και όσους έρχονται στην ώρα τους, αλλά να τους ανταμείβουμε. Σας καλωσορίζω λοιπόν, Αγκάρδια, και πάμε στο σημείο 11 της ημερική διάταξης, περιπολογισμός 2010, τμήμα 3. βεβαίω μπορούμε, όπως μου λένε εδώ πέρα, να τα δούμε και τα τρία σημεία ταυτόχρονα. τα τρία τμήματα του προϋπολογισμού. Λένα Εκ, ποιος... Οπότε δίνω τον λόγο στην συνάδελφο την κυρία Εκ για να μας πει πώς έχουν τα πράγματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα σύντομα να πω λίγα πράγματα για την έκθεσή μου για τον προϋπολογισμό. Πρώτα απ' όλα ζητώ συγγνώμη για το πολύ πιεσμένο πρόγραμμα, αλλά δεν οφείλεται αυτό στην Επιτροπή μας γιατί η ψηφοφορία είναι τον Οκτώβριο και συμπίπτει με ημερομηνίες της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμού και αν θέλαμε η δική μας ε, η γνώμη να ληφθεί υπόψη ε, έπρεπε να είναι τόσο πιεσμένο το πρόγραμμα και Συμφωνήσαμε έτσι στο πρόγραμμα αυτό με όλους τους συντονιστές πριν από τις διακοπές. Πρώτα απ' όλα αυτό. Γιατί κανονικά θα έπρεπε να είχαμε περισσότερο χρόνο για συζήτηση και για να μπορούν οι συνάδελφοι να τοποθετηθούν. Έχει επηρεάσει την δουλειά το πιεσμένο πρόγραμμα. Ναι και όχι. Είχαμε πολλές τροπολογίες από τις άλλες ομάδες και οι συνάδελφοι που ήταν εδώ και στην τελευταία θητεία βεβαίως γνωρίζουν τη διαδικασία. Και έχουμε και την στήριξη όλων σχεδόν των ομάδων, οπότε πρόκειται για μια έκθεση συνενετική όταν μιλάμε για την πολιτική έρευνας ε, και τεχνολογίας είναι κοινή τοποθέτηση της Επιτροπής. Τώρα οι στόχοι της ε, Επιτροπής είναι φιλόδοξοι όσον αφορά την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην ενέργεια, την, τον, την κοινωνία της πληροφορίας, την έρευνα και την τεχνολογία και την καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής και τη δημιουργία μιας οικοαποτελεσματικής οικονομίας, πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για εμάς Αλλιώς βεβαίω δεν θα ήμασταν και μέλη αυτής της Επιτροπής. Δυστυχώς το Συμβούλιο έκοψε τον προπολογισμό για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, που είναι το Ευρωπαϊκό Κοινό Ερευνητικό Πρόγραμμα, κατά 6% και 59% σε συγκεκριμένες γραμμές του προπολογισμού. Και η άποψή μου είναι και ελπίζω να συμφωνήσετε πως έτσι θα υπονομευθούν οι στόχοι της στρατηγικής της ε, Λισαβόνας για την ανάπτυξη δηλαδή ολόκληρης της εσωτερικής αγοράς. Οπότε, για να έχει Κομισιόν επαρκή προϋπολογισμό για να ασκήσει αυτή την πολιτική, θα πρέπει η Επιτροπή μας να στείλει ένα μήνυμα στην Επιτροπή Προπολογισμού πως ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποκατασταθούν οι αρχικές προτάσεις της ε, Κομισιόν και αυτό είναι και το βασικό μήνυμα της έκθεσης. Στο σχέδιο γνωμοδότησης που συζητάμε σήμερα προσπάθησα να συνοψίσω τα βασικά σημεία που είναι σημαντικά για την Επιτροπή μας. Προσπάθησα να ακολουθήσω αυτή τη γραμμή και στις ε, τροπολογίες που θα ψηφίσουμε και κατά βάση επαναφέρουμε τις ε, γράμμα σε αυτές τους προπολογισμούς στο αρχικό τους ύψος και χαίρομαι που οι συντονιστές είπαν πως θα υποστηρίξουν όλες σχεδόν τις τροπολογίες. Επίσης, υποστηρίζω κάποιες ιδέες και τροπολογίες των πρασίνων, αλλά αποφάσισα να μην τις υποστηρίξω όλες, γιατί θα ήθελα να δώσω μια κάποια ευελιξία στην Κομισιόν. Έχουμε μια γενική άποψη για το τι θέλουμε, αλλά το να τους δεσμεύσουμε τόσο δεν είναι και αποτελεσματικό. Τους δένουμε τα χέρια. Οπότε τους δίνουμε μια εντολή, θα αξιολογούμε τακτικά το τι γίνεται. Αλλά τώρα το να πούμε ακριβώς πού θα ξοδευτούν αυτά τα χρήματα δεν είναι σωστό. Δεν πρέπει να διεργούμε μεγαλύτερο διοικητικό άχθος από το απαραίτητο. Υποστηρίζω όμως συμβιβαστική λύση 1 καθώς η δημιουργία ενός υπερδικτύου είναι πράγματι απαραίτητη και το έλεγαν και αρκετές εκθέσεις πέρυσι. Οπότε υπάρχει και κάποια ευελιξία για την Κομισιόν. Τώρα οι τροπολογίες για την πυρηνική ενέργεια. Νομίζω πως η Κομισιόν θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να κάνει έρευνα. Έχουμε στην Επιτροπή ανθρώπους που αγαπούν την πυρηνική ενέργεια, άλλους που την αντιπαθούν και άλλους που την αντιπαθούν εντονότατα. Αυτό το οποίο έχουμε κοινό είναι ανεξαρτήτως της άποψής μας για την ποινική ενέργεια είναι πως η έρευνα είναι σημαντική, η ασφάλεια είναι σημαντική. Εάν ακολουθούσαμε λοιπόν τις τροπολογίες των πρασίνων δεν θα ήταν δυνατόν να έχουμε καμία ευρωπαϊκή έρευνα. Και παρά το ότι και εγώ δεν είμαι ένθερμη υποστηρικτής της ε, ποινικής ενέργειας, η έρευνα είναι πολύ σημαντική. Θέλω να τονίσω πως επαφίεται στα κράτη-μέλη το να αποφασίσουν αν θα έχουν πυρηνικού σταθμού στην ε, επικράτειά τους ή όχι. Το ενεργειακό μείγμα είναι τελείως εθνική υπόθεση. Εδώ μιλάμε για την ευρωπαϊκή έρευνα. Η έρευνα και η ασφάλεια έχει τεράστια σημασία για όλους μας καθώς έχουμε πυρηνικές εγκαταστάσεις στα μισά κράτη-μέλη. Με ναι, αυτή τη σύντομη παρουσίαση λοιπόν τελείωσα αναμένω τη συζήτηση με ενδιαφέρον και τις απόψεις των συναδέλφων και ελπίζω να έχουμε καλή ψηφοφορία στις 10. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή και για τη δουλειά σας τις τελευταίες ημέρες. Εσείς δουλεύατε ενώ οι άλλοι κάναν διακοπές. Το ίδιο ισχύει και για τους σκιώδεις συγητές που θα λάβουν τώρα το λόγο. Πρώτα απ' όλα η κυρία Ριέρα Μαδουρέλ. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για την πολύ καλή δουλειά της παρόλο που έκανε κούρσα κατά του χρόνου. Για τις τροπολογίες μας θα ήθελα να πω ότι η τροπολογία της ομάδος μου των σοσιαλιστών και δημοκρατών ως στόχο έχουν να ελαχιστοποιήσουν τις περικοπές του προϋπολογισμού τόσο στην έργεια όσο στην έρευνα και καινοτομία εφόσον, πράγμα που έχουμε πει πολλές φορές ε, σε αυτή την Επιτροπή, και η έρευνα και η καινοτομία είναι δύο απαραίτητοι πυλώνες στους οποίους πρέπει να βασιστούμε για να εξέλθουμε της κρίσεως. Επίσης, η ανάκτηση, η οικονομική ανάκτηση, θα είναι καρπός σε μεγάλο βαθμό αλλαγής του ενεργειακού μοντέλου που χρησιμοποιούμε μια πράσινη οικονομία, μια ενεργειακή αποταμίευση, η χρήση ανακυκλώσιμων πηγών ενεργείας, όλα αυτά είναι επιταγές. Οπότε δεν έχουμε την πολυτελή να περικόψουμε τον προϋπολογισμό. Εξάλλου η ατμομηχανή της ανάπτυξης ήταν πάντα η καινοτομία, η έρευνα και εξάλλου το πρόγραμμα ανάκαμψης του Προέδρου Ομπάμα το αναγνωρίζει αυτό εφόσον αύξησε σημαντικά τον προπολογισμό για την έρευνα. Στη θεωρία συμφωνούμε, αλλά στην πράξη η έρευνα και η καινοτομία υπαναχωρεί. Γι' αυτό θεωρώ ότι οι δύο αυτές γραμμές του προπολογισμού θα πρέπει να είναι ώστε να τον α, πλουσιότερες και επαναλαμβάνω, στόχος των τροπολογιών μας είναι να μειωθούν στο ελάχιστο οι περικοπές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Λάμπερτς κατόπιν. Do you hear me? Uh, so, well, first of all, uh, thank you. Πρώτα απ' όλα λοιπόν ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Εκ ε, για την ε, παρουσίαση του προπολογισμού που δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα εύκολο. Θα ήθελα να απαντήσω σε αυτά που είπατε για την πυρηνική ενέργεια και τις, τα σχόλια τα, τα πράσινα. Κοιτάξτε, αν δει κανεί την ιστορία και το πώς ακριβώς διαμορφώθηκε ο προπολογισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς πιστεύουμε ότι η πυρηνική ενέργεια υπερισχύει το θέμα δεν είναι ότι πρόκειται πλέον για τον ε, φτωχό αδελφό που ήταν ξεχασμένος εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή είναι θέμα πού ακριβώς στρέφει κανείς την προσοχή του. Οι πόροι είναι φιδωλοί, αυτό είναι αδιαμφισβήτο και δεν μπορούμε να τους επιμερίσουμε σε τόσα θέματα και σε τόσες πρωτοβουλίες. Όπως είπε και η Λένα, η πυρηνική ενέργεια είναι καθαρά θέμα των κρατών μελών. Εάν η Γαλλία επιθυμεί την πυρηνική ενέργεια, μπορεί κάλλιστα να δαπανεί τα δικά της κονδύλια, δεν χρειάζεται αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν εμείς καλούμεθα να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτό αυτό που μπορεί να κάνει τη διαφορά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτήν ε, λοιπόν την Επιτροπή και αλλού μιλήσαμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για την ε, μετατροπή της υποδομής, για το υπερδίκτυο, όλα αυτά που είναι σημαντικά. Η πυρηνική ενέργεια, εξάλλου, όπως την παρουσιάζουμε, δεν είναι απολύτως απαραίτητη. Και μην ξεχνάμε ότι η ποινική ενέργεια σίγουρα δεν βρίσκεται σε στενοπό. Αυτό λοιπόν είναι το αίτιο το οποίο μας οδήγησε στο να καταθέσουμε τις δικές μας τις προτάσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ρούμπιχ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω το Προεδρείο γιατί πράγματι δεν ήταν εύκολο ε, κατά τη διάρκεια των ε, διακοπών να διαδραματίσει κανεί το ρόλο του συντονιστή και νομίζω οι συντονιστές ε, εργάστηκαν θαυμάσια γιατί δεν είναι αυτονόητο ότι έγκαιρα θα μπορεί κανείς να εμφανιστεί με αποτέλεσμα ψηφοφορίας ως Επιτροπή. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστώ ιδιαίτερα θερμά. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι Λόγω της οικονομικής κρίσης και της ενεργειακής ασφάλειας πρέπει να παίξουμε σημαντικό ρόλο, να προχωρήσει η χρηματοδότηση. Το πρόγραμμα SIPT ε, σχετικά με τις καινοτομίες είναι πολύ σημαντικό, κυρίως για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να προωθήσουμε την ασφάλεια των θέσεων εργασίας. Και το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, το οποίο πλέον θα αποκτήσει μια διαφορετική έμφαση το πρόγραμμα αυτό πρέπει να το φέρουμε στο επίκεντρο των προσπαθειών μας. Και εγώ ε, στηρίζω αυτή την τροπολογία των πρασίων για τα ε, διευρωπαϊκά δίκτυα. Όπως ακούσαμε χθε, αν θέλει κανείς να χρησιμοποιήσει την ε, ολική ενέργεια ε, δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει ένα αποτελεσματικό δίκτυο στην Ευρώπη. Και γι' αυτό ε, θεωρώ ότι είναι καθοριστική σημασία η πρόταση η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιληφθεί των διευρωπαϊκών δικτύων κυρίως στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Και εμείς πρέπει να αναλάβουμε την πρωτοβουλία έτσι ώστε τα δίκτυα αυτά να συσταθούν το συντομότερο δυνατόν. Το τρίτο που θέλω να πω είναι η αποκαλούμενη ευφύης ενέργεια. Εμείς επιθυμούμε να υπάρχει ευελιξία στη χρήση και βεβαίως και η πυρηνική ενέργεια συζητήθηκε στη δική μας πολιτική ομάδα όπου δίστανται οι απόψεις. Εκεί όμως που συμφωνούμε όλοι είναι ότι η ασφάλεια πρέπει να προβάλλεται πάνω απ' όλα είναι απαραίτητο να υπάρξει κάποια επανεξέταση του θέματος έτσι ώστε να προσφέρουμε τη διαφάνεια στην ασφάλεια. Εξάλλου να πω ότι η δική μας Επιτροπή οφείλει να προσπαθήσει τις απόψεις μας να τις περάσει στην Ολομέλεια. Εδώ λοιπόν καλώ την εισηγήτρια να έχουμε μια στενή συνεργασία με την Επιτροπή των Προπολογισμών, να ε, συνεργαστούμε με τους αρμόδιους, έτσι ώστε οι αποφάσεις να μην είναι ατομικές, αλλά να αποφασίσουμε ως Επιτροπή και αυτές οι αποφάσεις μας να εμφανιστούν στους καταλόγους ψηφοφορίας. Επόμενος ε, δεν είμαι σίγουρος αν πρόφερα καλά το όνομά σας. Κύριε Πρόεδρε, Αυτά είναι τα πρώτα βήματα που γίνονται για μας. Δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν οι εργασίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, τα ε, παλαιά μέλη της Επιτροπής για την ε, εργασία τους, σε σχετικά με τη χρηματοδότηση σημαντικών προγραμμάτων. Όλοι μας συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνουν επενδύσεις στην υποδομή, στις νέες διασυνδέσεις, έτσι ώστε να μην καταλήξουμε με ενεργειακές νησίδες, όπως συμβαίνει με την περίπτωση της Βαλτικής. Υπάρχουν και άλλες παρεμφερείς περιπτώσεις. Αυτό που θέλω να προβάλλω είναι ότι πρέπει να υπάρχει ασφάλεια στην πυρηνική ενέργεια η ανακύκλωση των πυρηνικών καταλήπων, όπως επίσης και η πάυση λειτουργίας των ε, αντιδραστήρων, είναι θέματα που χρήζουν ιδιαίτερη προσοχή. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η δική μας ε, ε, πολιτική ομάδα θα στηρίξει αυτές όλες τις τροπολογίες που κατατέθηκαν. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μπάλσο. Αγαπητοί συνάδελφοι, κοιτάξτε, είναι μεγάλη ευθύνη αυτή που αναλαμβάνει κανείς ε, ως ε, νεοεκλογής ε, ευρωβουλευτής να λάβει το λόγο. Το δικό μου το κόμμα μέχρι τώρα δεν είχε εκπροσώπηση στην Επιτροπή σας. Αντί όμως ε, να σιωπήσω, προτίμησα να λάβω το λόγο. Για τον εξή λόγο διότι υπάρχει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και θα ήθελα να επιβεβαιώσω αυτά τα οποία είπε η κυρία εισηγήτρια. Στηρίζω την ε, ισόρροπη θέση της, ε, κυρίως όσον αφορά τους πόρους που θα πρέπει να προβλεφθούν για την ενέργεια και την έρευνα, με για την έρευνα. Κυρίως έρευνα για την πυρηνική ενέργεια, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το θέμα δεν είναι κατά πόσον θα ε, κατασκευαστούν πυρηνικοί αντιδραστήρες. Αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι θα πρέπει να δράσουμε έχοντας κυρίως κατά νου την ασφάλεια των πυρηνικών αντιδραστήρων. Αυτός είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ λοιπόν δεν θεωρώ ότι αυτό ε, αφορά ένα και μόνο κράτος μέλος ότι αναπόκειται στη δική του τη διακριτική ευχαίρεια να αποφασίσει όχι. Όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια, ε, όλοι φέρουμε ευθύνη για το μέλλον. Βεβαίως και τα σώμεθα υπέρ της ε, πράσινης ενέργειας, θέλουμε να επιτύχουμε, να φτάσουμε σε τέτοιο τεχνολογικό επίπεδο, έτσι ώστε να μην χρειάζεται καν να κάνουμε αυτή τη συζήτηση μετά από 20 χρόνια. Αν όμως έχει κανείς κατά νου την κλιματική αλλαγή, τις ε, εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα, ε, οφείλει να ομολογήσει ότι η πυρηνική ενέργεια είναι καθαρή ενέργεια. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι εμείς ε, συμφωνούμε με την ισορροπία που χαρακτηρίζει την ε, ε, παρουσίαση της ομιλήτριας Και επανέρχομαι τώρα στους καταναλωτές. Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, το ύψος των τιμών είναι αποδεκτό για τους πολίτες μόνο εφόσον και η πυρηνική ενέργεια καταλαμβάνει τον ρόλο που τη αξίζει και α μην ξεχνάμε ότι αυτή είναι και η φτηνότερη πηγή ενέργεια. Κυρία Εκ, θέλετε εσεί να πείτε κάτι ή δεν ξέρω, υπάρχει κάποιο από την Κομισιόν που θέλει να λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρετε, Φιλίπε ονομάζομαι και εκπροσωπώ τη ΓΑΜΑ Ενέργειας και Μεταφορών. Τα σχόλιά μου αφορούν μόνο την ε, γραμμή του προπολογισμού 06. Θα θέλαμε εκ μέρους της Γενικής μας Διεύθυνσης να σας ευχαριστήσουμε την Επιτροπή σας και την εισηγήτριά σας που τοποθετηθήκατε σε σχέση με το σχέδιο προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τρία σχόλια για την 6101 και 6109 τροπολογίες που προτείνουν αύξηση των ε, κονδυλίων 1 εκατομμύριο για την ενεργειακή πολιτική και 5 εκατομμύρια για την έρευνα που αφορά την ενέργεια. Εμείς έχουμε την άποψη ότι αυτές οι αυξήσεις δεν χρειάζονται δεδομένης της ε, κατάστασης ε, που αφορά την εφαρμογή του τρέχοντος προγράμματος. Μιλώ για τις πληρωμές και όχι για τις ε, δεσμεύσεις πληρωμών. Για την 6178 συμφωνούμε, όπως και για την 6179 για τη λεγόμενη ΕΦΗ ενέργεια e και το σχετικό πρόγραμμα. Έχουμε όμως την άποψη ότι η προτινόμενη αύξηση για αυτή την τελευταία ε, τροπολογία 87 εκατομμύρια 8,7 ε, μάλλον 18,7 ε, είναι υπερβολικό 10 είναι αρκετά πιστεύουμε και ομιλώ αποκλειστικά και πάλι για τις αυξήσεις ό,τι αφορά τις πληρωμές και όχι τις υποχρεώσεις για την 6173 για τα ενεργειακά προγράμματα που θα βοηθήσουν στην οικονομική ανάκαμψη. Θέλουμε να προτείνουμε την προσθήκη ενός κειμένου. Θέλετε να προσθεθεί ένα κείμενο το οποίο είναι συγγενές με το δικό μας, αλλά το if appropriate, όπου δει αν είναι κατάλληλο, διαγράφεται, ε, οπότε θεωρούμε ότι αφού παραθέτεται, γιατί ουσιαστικά περί αυτού πρόκειται, αφού αναφέρεται αν θέλετε ένα κείμενο τη Κομισιόν, θα πρέπει να παρατήσετε αυτούσιο και όχι αλλοιωμένο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η συνάδελφο η κυρία Εκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα έχουμε τριπλή κρίση. Βεβαίως την χρήματο-οικονομική που θα επιληθεί μια κρίση θέσεων εργασίας και μια κλιματική κρίση. Για να λυθεί αυτό, να λυθούν όλα αυτά, οι ευθύνες που έχουμε στην ε, Επιτροπή μας είναι κορυφαία σημασία. Η πολιτική βιομηχανία, έρευνα, ο τομέας της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών είναι πολύ σημαντικά εργαλεία και βρισκόμαστε σε μια συζήτηση για τον προϋπολογισμό και είμαστε σε ανταγωνισμό με όλες τις άλλες επιτροπές και τις πολιτικές τους ευθύνες. Οπότε αυτό το οποίο προσπάθησα να κάνω είναι πρώτα απ' όλα να μην έχω μια πολύ αναλυτική έκθεση, αλλά μια μικρή και επικεντρωμένη για να είναι σαφείς οι προτεραιότητές μας, να μην υπάρχει αμφιβολία στους συναδέλφους της ε, Επιτροπής ε, Προπολογισμού για το ποιες είναι οι προτεραιότητές μας. Για να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που έχουμε για να λύσουμε αυτή την τριπλή κρίση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και ο κόσμος. Γι' αυτό έχουμε αυτούς τους ε, στόχους. Επίσης, οι συνάδελφοι θεωρούν, εάν δείτε όλες τις ε, τροπολογίες που έχουν κατατεθεί από όλες τις ομάδες, θα δείτε πως ε, έχουν ε, τις ίδιες ακριβώς ανησυχίες, γι' αυτό και έχουμε επικεντρωθεί σε αυτά τα 8 σημεία. Βεβαίως, θα έχουμε πάρα πολλά παζαρέματα στην Επιτροπή Προϋπολογισμού και ελπίζω να έχουμε πλειοψηφία για τον κατάλογο ψηφοφορία που προτείνω και μετά να τον συζητήσουμε και στις όταν θα το συζητήσουμε στις πολιτικές μας ομάδες, να υποστηρίξετε αυτούς τους τομείς που περιέχει η έκθεση. Αυτό εδώ δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή της συζήτησης του προπολογισμού, οπότε δεν ανησυχώ ιδιαίτερα για το να έχουμε λίγα περισσότερα εκατομμύρια από αυτά που θέλει η Κομισιόν στο τέλος. Γιατί, πιστέψτε με, θα δοθεί αγώνας για κάθε ευρώ του προπολογισμού και στους τομείς αυτούς θα ήθελα να υπενθυμίσω την συζήτηση που είχαμε με Συμβούλιο και Κομισιόν και ειδικά με το Συμβούλιο για ολόκληρη την δημοσιονομική περίοδο όταν ξεκίνησε το Συμβούλιο με το να κόψει τη χρηματοδότηση της έρευνας κατά 5%. Καταστροφή δηλαδή για την έρευνα και την καινοτομία. Και η τελική μάχη ήταν τόσο σκληρή ώστε λίγες εβδομάδε πριν ξεκινήσει το δημοσιονομικό έτος δεν είχαμε λάβει απόφαση. Οπότε ήμασταν σχεδόν έτοιμοι να καταφύγουμε σε μια θέση παναχώρηση, να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή τον προπολογισμό του προηγούμενου έτους. Οπότε θα είναι δύσκολες συζητήσεις, πρέπει να είμαστε πολύ επικεντρωμένοι στην έκθεση και στον κατάλογο σοφορίες και ο συνάδελφος ο κ. Ρουβιχέ τα ξέρει αυτά, ξέρει τι μάχη είχαμε δώσει. Οπότε θα ήθελα να ευχαριστήσω τους και οδησηγητές και όσους μίλησαν για την υποστήριξή τους και θα ήθελα να ζητήσω την ε, στήριξή σας ε, εντός των πολιτικών ομάδων σας γιατί βεβαίως θα συζητηθούν όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την διευκρίνηση καθώς που δεν είναι σημαντική μόνο για την Επιτροπή μας αλλά και για το τι θα κάνουμε στις ομάδες γιατί βεβαίως στο τέλος ε, η Επιτροπή Προπολογισμού είναι αυτή που θα παίξει τον βασικό ρόλο και σας ευχαριστώ που ξεκαθαρίσετε ότι μόλις τώρα αρχίζει η δουλειά μας. Καλό είναι να το έχουμε αυτό κατά νου γιατί μετά θα πρέπει ο καθένας να πάει στην κοινοβουλευτική του ομάδα και να ασκήσει κατάλληλες Δεν βλέπω κανέναν να ζητάει τον λόγο οπότε περνάμε να σας υπενθυμίσω στο σημείο 11 πως ε, αυτή τη στιγμή μόνο το συζητάμε. 8 Σεπτεμβρίου 12 η ώρα είναι η προθεσμία για τροπολογίες. Οπότε 29 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή και ο προϋπολογισμός ε, το σχετικό ψήφισμα θα εγκριθεί στις 8 Οκτωβρίου. Δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση. Οπότε έτσι θα γίνει. Μετά περνάμε στο σημείο 12 που είναι οι συγκεκριμένες τροπολογίες. Να υπενθυμίσω πως έχουμε 84 τροπολογίες που έχουν συζητηθεί. Οπότε θα τις δούμε από κοινού. Νομίζω πως είναι μεταφρασμένες και σε όλες τις ε, γλώσσες έτσι ώστε να μπορέσουμε σήμερα όχι μόνο να συζητήσουμε αλλά να ψηφίσουμε κιόλας. έτσι ώστε να είμαστε εντός των προθεσμιών, ώστε στις 9 Σεπτεμβρίου να υποβάλουμε και τα δικά μας έγγραφα. 28 και 29 Σεπτεμβρίου, Ολομέλεια. Ξεκάθαρα και αυτά, οπότε μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 13, η ψηφοφορία, αλλά δυστυχώς διαπιστώνω εδώ πως πρέπει να ξεκινήσει στις 10 η ώρα. Οπότε ε, κερδίσαμε και λίγο χρόνο. Οπότε θα κάνουμε ένα διαλυματάκι, πιείτε ένα καφέ, αλλά παρακαλώ ακριβώς 10 η ώρα, να είστε σίγουροι 10 η ώρα θα ξεκινήσει η ψηφοφορία. Για να συνηθίζουμε και όλα, θα ξεκινάμε στην ώρα μας, θα κερδίσουμε πολύ χρόνο τους επόμενους μήνες. Λοιπόν, 10 η ώρα ακριβώς ξεκινάμε. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση όπως σας υποσχέθηκα ή σα απείλησα μάλλον. Ξεκινάμε ακριβώς την ώρα μας. Ελπίζω να έχετε τις κάρτες για την ψηφοφορία. Μπορεί να τις χρειαστούμε, ελπίζω όχι, αλλά μπορεί. Θα προσπαθήσουμε πρώτα απ' όλα χωρίς τις κάρτες. Να δούμε. Κοιτάξτε, βουλευτές χωρίς κάρτα δεν είναι βουλευτές. Ε, εννοώ για τις ε, ψηφοφορίες, έτσι. Λοιπόν. Έχουμε 84 τροπολογίες. Έχετε τον κατάλογο ψηφοφοριών, ελπίζω όλοι, για να ξεκινήσουμε. να κάνουμε μια δοκιμή με την κάρτα μέχρι να έρθουν και όλοι στην αίθουσα. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Ψηφίζω τώρα για το εάν θα συνεδριάσουμε και αύριο. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεν δουλεύει.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 και το 46 εκεί δεν δουλεύει νομίζω. Κάποιες ε, μηχανές δεν δουλεύουν γιατί είναι πολύ νέα η Εύσα και τα μηχανήματα ούτε το δικό σας. Ε, τεχνολογία και Λάμπερτς ούτε το δικό σας λειτουργεί εξακολουθεί να είναι ανοιχτή ακόμα η ψηφοφορία. Πατήστε γερά το κουμπάκι. Πρέπει να, να μας βοηθήσουμε για να δούμε. Ε, να δοκιμάσω κάπου αλλού. Problem. Λάμπερτς, δουλεύει τώρα, όχι. Funktioniert nicht. Uh, some machines don't work. I think so. Κάποια μηχανήματα δεν δουλεύουν. <laughs> Gibt es noch eine Maschine, die nicht funktioniert? Υπάρχει κάποιο μηχάνημα που δεν δουλεύει ακόμα. Ακόμα. Ακόμα δεν δουλεύει. Ε, Έπρεπε να μας βοηθήσει ο τεχνικός εδώ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 Δουλεύει τώρα. Ωραία. Κάποιος άλλος έχει προβλήματα ακόμα. Αν είναι καθίστε αλλού. Έτοιμοι. Τελείωσε λοιπόν αυτή η ψηφοφορία. Το αποτέλεσμα είναι 41 υπέρ, 20, ε, 41 ψήφισαν όχι, 22 υπέρ, 13 κατά, 6 αποχές. Συν Δύο ακόμα υπέρ. 24 υπέρ. Αποφασίστε λοιπόν ότι αύριο θα συνεδριάσουμε. Ε, εντάξει, τους άλλους δοκιμή ήταν μόνο. Λοιπόν, πρώτη τροπολογία. Τούρμες. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Όχι, διανατάσεως της χειρός. Νομίζω Διανατάσεις χειρός και θα μετρήσουμε και στην... Λοιπόν, πρώτη τροπολογία 02, 01, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το νου... ίδιο νούμερο 02 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 04 υπέρ Ευχαριστώ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 0430 υπέρ. Κατά. Αποχές. Κανείς ένας εγκρίνεται. 501 υπέρ. Κατά. Αποχές. Μία εγκρίνεται. 503 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 201 61.00 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται οπότε 61-40 κατά πίπτη. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ορίστε. Eh, eh, Υπάρχει κάποια σύγχυση και δεν μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε. Λοιπόν, θα κάνουμε το εξής θα λέω πάντα το νούμερο της τροπολογίας της δικής μας επιτροπή, είναι, της ε, επιτροπής. Οπότε η 6140 τελειώσαμε. Ναι, ναι, ευχαριστώ για την υπόδειξη. 6141 υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6142 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6143 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 61-44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 07 άρα εγκρίνεται και αυτή 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61-77 καταπίπτει 61-08 υπέρ κατά αποχές μία εγκρίνεται 61-46 πέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61-47 υπέρ κατά αποχές 6178 61-78 αποσύρεται 61-48 υπέρ κατά αποχές μία εγκρίνεται 61-49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61-50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61-51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Περνάμε συμβαστική λύση 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οπότε οι 61, 61 και 61, 71 φεύγουν. Οπότε πάμε στην 61, 55 υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61, 01 υπέρ. Κατά. αποχές εγκρίνεται 61-52 υπέρ Α, με συγχωρείτε απορρίπτεται 61-52 έχει αποσυρθεί ε, συμβα... συμβαστική λύση 2 υπέρ ναι πρέπει να μετρήσουμε Όχι, όχι. Καλύτερα με το διανατάσεις χειρό. Gegenstimmen. Κατά. Αποχές. απορρίπτεται με 22 εναντί 32 και 2 αποχές. Οπότε έχουμε την 61 6102. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Εγκρίνεται. Αποχές. Εγκρίνεται. 61. Όχι. Καταπίπτει. 75. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 6173 61-73 υπέρ. Κατά. Αποχές. απορριπτεται 61.84 61-84 υπέρ. Κατά. Αποχές. Κάποιες ψηφικατά, κατά εγκρίνεται. 6109 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 6176 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 6156 Μάλιστα καταπίπτει. 61-54 υπέρ κατά αποχές ευχαριστώ εγκρίνεται 61-10 οπότε καταπίπτει 61-60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61-58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61-59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61-57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61-62 υπέρ κατά αποχές ομόφωνα όχι με μία αποχή 61-63 υπέρ κατά αποχές ομόφωνα 61-64 υπέρ κατά αποχές μία εγκρίνεται 61-65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61-04 και 61-66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61.05 και 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61.12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61.23 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 61-32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61-13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61-33 υπέρ. 33, ναι. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μπορούμε να ψησουμε καποιες κάποιες μαζί. Όχι. Εντάξει. 61-24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61-21 υπέρ. Ναι. Όχι. Ε, κατά. Αποχές. 61-22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61-20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61-31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61-83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61-11 και 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 να επαναλάβω ε, σε αυτή τη σελίδα μπορούμε να κάνουμε μια ομαδική ψηφοφορία να ψήσουμε όλη τη σελίδα μαζί από την 61 30 μέχρι την 14 61-14. Όποιος είναι υπέρ όλων αυτών, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Οπότε από την 61-30 μέχρι την 61-14 εγκρίνονται 61-81 υπέρ. Ευχαριστώ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61-69 καταπίπτει. Ευχαριστώ. 61-80 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61-74 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61-68 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Αυτό ήταν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, γρήγορη αυτή ψηφοφορία. Έχουμε βεβαίω και την συνολική ψηφοφορία στο τέλος. Ποιος ψηφίζει λοιπόν το συνολικό πακέτο όπως ε, έχει διαμορφωθεί. Παρακαλώ ηλεκτρονικά και όσοι συνάδελφοι δεν έχουν κάρτα θα τους μετρήσουμε ξεχωριστά. Πρώτα απ' όλα λοιπόν ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Είναι τρεις παραπάνω από το ΕΛΚ και ένα σοσιαλδημοκράτης παραπάνω. Παρακαλώ προσεκτικά βγάλτε τις καρτούλες σας. Sind wir klar? Noch nicht? Ε, εντάξει, όλα εντάξει, οπότε λίγη ψηφοφορία. Υπάρχει κάποιος που δεν μπόρεσε να ψηφίσει και πρέπει να ψηφίσει χωρίς κάρτα. Άλλη μία αποχή λοιπόν. Μία αποχή ακόμα. 48 Abstimmung, 43 dafür,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 Liebe Kolleginnen, liebe Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ξανακαλωσορίζω, χαίρομαι που είσαστε όλοι εδώ. Εν τω μεταξύ έχει έρθει ο προσκεκλημένος μας και αν και έτυχε και δεν το προσέξατε, γιατί έχει και πολύ θόρυβο μέσα στην αίθουσα, Αγαπητοί συνάδελφοι, έχετε την καλοσύνη, αν θέλετε να έχετε κατηδίαν συζητήσεις, να εγκαταλείψετε την αίθουσα. Γιατί έχουμε έναν ε, καλεσμένο και νομίζω ότι σωστό είναι να είμαστε ίσχυοι και να ε, προσέξουμε αυτά που θα πει. Τον καλωσορίζω λοιπόν τον προσκεκλημένο μας, ε, τον κύριο Τομπίας Κραντς, ο οποίος είναι Υπουργός Ανώτερης Εκπαίδευσης και Έρευνας, Προεδρεύων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Κραντς, Έχετε πρόβλημα. Κύριε Κράντς, λοιπόν, χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήρθατε. Εχθές ε, ήδη δεχθήκαμε δύο συναδέλφους σας και πρέπει να σας πω ότι περιμένουμε με αγωνία αυτά τα οποία θα μας πείτε. Θα ήθελα ε, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, να σας δώσω το λόγο. Θα ήθελα τους αντέλφους ε, να σας αφιερώσουν την προσοχή τους και μετά, αν δεν έχετε αντίρρηση, θα θέλαμε να συζητήσουμε μαζί σας. Και άλλη μια φορά καλωσορίσατε και έχετε το λόγο. Herr ordförande, eh, av Europaparlamentet αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. <clears throat> Πρέπει να σας πω ότι είναι μεγάλη χαρά για μένα το ότι ε, μπορώ να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Ουδικής Προεδρίας ε, στον ε, τομέα της έρευνας. Είμαστε λοιπόν ευγνώμονες στην προηγούμενη Προεδρία για το έργο που παρουσίασε η Σουηδική Προεδρία εμφανίζεται, αναλαμβάνει σε κάποια στιγμή, όπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκύπτουν σημαντικέ προκλήσει. Βρισκόμαστε μεσούσει ε, τη μεγαλύτερη παγκόσμια οικονομική κρίση από τη δεκαετία του 30. Η ε, γρήπη των χείρων όλο και περισσότερο διαδίδεται και η κλιματική απειλή επίσης καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική. Έτσι λοιπόν ε, πλέον καλούμεθα να δράσουμε. Στην ε, Σουηδία οι Υπουργοί έχουν ε, συνειδητοποιήσει την σημασία όλων αυτών των προβλημάτων. Αυτή τη στιγμή η επενδύσεις που κάνουμε στην έρευνα αποτελούν τον πυλώνα των προσπαθειών μας. Ε, πρέπει λοιπόν να λάβουμε όλες τις ευθύνες μας, να αγωνιστούμε για να διασφαλίσουμε ότι ε, θα έχουμε πράγματι στραμμένο το βλέμμα προς το μέλλον. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την έρευνα. Πολλές χώρες επενδύουν μεγάλα κονδύλια στην έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν πολλά φιλόδοξα προγράμματα. Η Σουηδική Προεδρία έχει επισημάνει αρκετές προτεραιότητε στον τομέα της έρευνα. πρώτα απ' όλα την διαχείριση του τομέα της Ευρωπαϊκής Έρευνα, κατόπιν το τρίγωνο τη της και τέλος το μέλλον για το ε, πρόγραμμα πλαίσιο. Όταν πρόκειται για το ERA, τον Ευρωπαϊκό ε, Χώρο Έρευνας, ε, πάντα θέλουμε την αποτελεσματικότητα, την προβολή και την ιεράρχηση. Η αποτελεσματικότητα σημαίνει σαφέστατη και σα... διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Χώρου. Η Σουηδία πιστεύει ότι ένα μεγάλο τμήμα των κονδυλίων τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κατευθύνονται στην καινοτομία, την ε, έρευνα και σε άλλα μέτρα που προάγουν την ανταγωνιστικότητα. Πιστεύω όμω επίση ότι οι πόροι που τώρα κατευθύνονται στην έρευνα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικότερα. Είναι απαραίτητο να υπάρχει συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο, χωρί βεβαίω να θέτει κανεί σε κίνδυνο την πολυμορφία των προσεγγίσεων που και αυτή τη χρειαζόμαθα. Πολλά μέτρα, η εργαλεία όπω εμεί τα αποκαλούμε, είναι υπόκεινται ε, στη διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών, συγκεκριμένων ομάδων στόχων και ειδικών προβλημάτων που καλούμεθα να λύσουμε. Αυτός εξάλλου και ο πλουραλισμός και η ισχυρή πλευρά της έρευνας ε, που καλούμεθα να υπηρετήσουμε. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να αυξήσουμε τα ωφέλη που προκύπτουν από τις επενδύσεις μας. Είναι λοιπόν ένα θέμα ε, του οποίου πρέπει να επιληφθούν τα κράτη-μέλη. Ο ευρωπαϊκός χώρος της έρευνας ε, πρέπει να είναι σαφέστερος. Οι πολίτες Ευρώπης πρέπει να βλέπουν ότι οι επενδύσεις στην έρευνα μπορούν πράγματι να προσφέρουν την ειδοποιώ διαφορά στην καθημερινή τους ζωή. Στις αρχές Ιουλίου η Προεδρία οργάνωσε ένα συνέδριο για το μέλλον της έρευνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το συνέδριο έλαβε χώρα στο Λαντ, στη Νότιο Σουηδία και τα αποτελέσματα του συνεδρίου είναι τώρα γνωστά ως η δήλωση του ΛΑΝΤ. Το συνέδριο επισήμανε ότι η έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να λαμβάνει όλο και περισσότερο υπόψη τη τι ε, προκλήσει που αντιμετωπίζουμε, την κλιματική αλλαγή, την πρόσβαση στα τρόφιμα, την ε, αηφόρο ε, ενέργεια, την διασφάλιση των υδάτινων πόρων και τις πανδημίες. Η δήλωση του Λούντ εξάλλου εξετάζει και το πόσα ακριβώς εντοπίζονται οι προτεραιότητες στην ευρωπαϊκή έρευνα. Μέχρι τώρα η Κομισιόν ήταν εκείνη που ασχολείται με τις προτεραιότητες, αυτό όμως πια δεν είναι αποδεκτό. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να είναι ανοιχτές και να συμπεριλαμβάνουν όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό χώρο. Εάν λοιπόν επιθυμούμε οι προσπάθειές μας να ευοδοθούν σε σχέση με τις ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, εμείς στο Συμβούλιο και εσείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να άγουμε τις διαδικασίες αυτές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα λοιπόν που συζητάμε για το πώς ακριβώς μπορεί να εξελιχθεί περιττέρω ο ευρωπαϊκός χώρος της έρευνας, το θέμα δεν είναι απλά να περιμένουμε τις προτάσεις της Κομισιόν. Πάρα πολλά ε, εναπόκεινται και στην κινητοποίηση των εθνικών και περιφερειακών αρχών και φορέων. Ε, είναι θέμα των θεσμών της κοινότητας, αλλά και πολλών άλλων της κοινωνίας των πολιτών, που όλοι αυτοί καλούνται να λειτουργήσουν μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο της έρευνας. Η συμμετοχή και η συζήτηση για το πώς θα διαμορφωθεί αυτή η συνεργασία είναι καθοριστική σημασία. Γι' αυτό το λόγο η Σουηδική Προεδρία οργανώνει ένα σεμινάριο σε υπουργικό επίπεδο στι 24 Σεπτεμβρίου, την ημέρα πριν λάβει χώρα το Συμβούλιο Υπουργών Έρευνα στο Συμβούλιο. Αυτό θα το διοργανώσουμε από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί θεωρούμε ότι από κοινού μπορούμε να ε, συμβάλλουμε καθοριστικά στα μελλοντικά προγράμματα. Το σεμινάριο θα εξετάσει θέματα όπως ε, τον κόσμο, το 2025 και θα κληθούμε λοιπόν ε, να στρέψουμε το μέλλον μας ε, σε ένα χρονικό διάστημα μετά από 15 χρόνια. Το να ενισχύσει κανείς την έρευνα δεν αρκεί για την παγκόσμια οικονομία, για να ανακάμψει. Η Σουηδική Προεδρία ε, προτίμησε να εραρχήσει κάποια θέματα που έχουν σχέση με το απακολούμενο τρίγωνο της γνώσης, δηλαδή την αλληλένδεση, την αλληλεξάρτηση ανάμεσα στην ανώτατη έρευνα, ανώτατη παιδεία, την έρευνα και την καινοτομία. Μόλις ήρθα από ένα συνέδριο στο και ένα συνέδριο που είχε σχέση με την έρευνα και την παιδεία. Και εκεί συζητήσαμε ακριβώς αυτά τα θέματα, την δύναμη της ε, καινοτομίας. Στη Σουηδία και γενικότερα στην Ευρώπη ε, έχουμε σημαντικές επενδύσεις στην έρευνα. Το θέμα όμως είναι ότι λίγα από τα αποτελέσματα της έρευνας ε, καθίστανται ε, αντικείμενο εμπορευματοποίησης. Υπάρχει λοιπόν ένα παράδοξο και αυτό πρέπει να το εξετάσουμε σε σχέση με την ευημερία μας. Η έρευνα βεβαίως και αξίζει χάρη αυτής και μόνο, αλλά πρέπει να αποφέρει και ωφέλη στην κοινωνία. Η τα αποτελέσματα της έρευνας στην ιατρική δεν μπορούν να παραμένουν στα ντουλάπια των εργαστηρίων, πρέπει να ωφελούν την κοινωνία και πρέπει να συζητήσουμε και το πώς μπορούν να εξυγχρονιστούν τα πανεπιστήμια για να λειτουργούν αποτελεσματικά και να είναι ανταγωνιστικά στην εποχή της, ε, ε, του ανταγωνισμού. Κάτι άλλο που θέλουμε να προβάλλουμε είναι η ποιότητα των πανεπιστημίων και άλλων ερευνητικών φορέων. Αυτό είναι εξίσου σημαντικό για να έχουμε ένα υγιές μέλλον. Πολύ λίγα πανεπιστήμια ευρωπαϊκά εμφανίζονται στις ε, λίστες αξιολόγηση Κατά την άποψή μα λοιπόν να υπάρξουν περισσότερε επενδύσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να στηρίξουμε του θεσμού αυτού τη Ευρωπαϊκή Γνώση. Κατά τη διάρκεια τη δική μα προεδρία, θα προτείνουμε συγκεκριμένη στρατηγική σε αυτόν τον τομέα. Και κατά τη διάρκεια τη προεδρία μα θέλουμε να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για το πρόγραμμα πλαίσιο και το μέλλον του. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό ε, να έχουμε φιλοδοξίε υψηλού επίπεδου όσον αφορά μόνο την ποιότητα αλλά και την αποτελεσματικότητα. Θεωρούμε τι στόχοι μας μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα αν είναι περισσότερο στρατηγικοί. Πρέπει να εξορθολογήσουμε του κείμενου κανονισμού, να αναζητήσουμε λύσει οι οποίε θα μα οδηγήσουν εκτό του πλαισίου που χρησιμοποιούμε σήμερα. Πιστεύω ότι πρέπει να απλουστεύσουμε το διοικητικό άχθο. που αντιμετωπίζει η έρευνα αναζητώντα κονδύλια. Όλοι μα οι Κομισιόν, τα κρατημέλη και το Κοινοβούλιο μπορούν να βοηθήσουν. Και ένα τρόπο για να ενισχύσουμε την ε, έρευνα είναι να υπάρχει πιο συγκεκριμένη συνεργασία ανάμεσα μέσα από κοινά προγράμματα. Είμαστε ακράδαντα ανταπεπισμένοι ότι από τον καλύτερο συντονισμό των διαφόρων εθνικών προγραμμάτων θα προκύψουν σημαντικά ωφέλη. Το Συμβούλιο ενέκνε τα αποτελέσματα και ε, έτσι λοιπόν καλούμεθα να αποφασίσουμε για την πρώτη σειρά προγραμμάτων που θα αρχίσουν να ισχύουν το 2010. Ξέρετε ότι υπάρχει μια ομάδα υψηλού επίπεδου που αυτή τη στιγμή δουλεύει σε συγκεκριμένε προτάσει και γνωρίζουμε καλά ότι θα επιτευχθεί πρόοδος ε, από, στην αντιμετώπιση των ασθενειών. Θέλουμε να καταθέσουμε ε, πρόταση για ε, έρευνα και πέρα από τη δική μας την Προεδρία. Τελειώνοντας, δεν θέλω να φέρω και ένα άλλο θέμα που ε, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Η στρατηγική μας για την Βαλτική. Αυτή είναι πρώτη προτεραιότητα για τη Σουηδική Προεδρία. Θέλουμε να υπάρχει συνεργασία με τις χώρες της Βαλτικής στον τομέα της έρευνας εδώ και χρόνια. Υπάρχει συνεργασία με τις χώρες της Βαλτικής για θέματα περιβάλλοντος ε, υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το πρόγραμμα Bonus ε, θα πρέπει να εγκριθεί με βάση το άρθρο 169. Έτσι λοιπόν η Κομισιόν ε, θα πρέπει να καταθέσει προτάσεις σε σχέση με το πρόγραμμα αυτό για να ληφθούν υπόψη. Ε, πρόεδρε, αγαπητά μέλη, έχουμε μια θαυμάσια αγαστή σχέση ανάμεσά μας ε, και αυτό πρέπει να υπάρχει και στο μέλλον. Είναι καθοριστική σημασία για την εφαρμογή του προγράμματος και γι' αυτό σας καλούμε να συνεχίσουμε την αγαστή συνεργασία που υπήρχε ανέκαθεν ανάμεσα στην Επιτροπή αυτή και το Συμβούλιο. Έτσι ώστε πράγματι να μπορέσουν οι πολίτες της Ευρώπης να ωφεληθούν. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο εφόσον υπάρχει συνεργασία ανάμεσα επιχειρήσει και την έρευνα. Σα συγχαίρω για την εκλογή σα ε, και ε, ελπίζω να μπορέσω να συναντήσω όσο δυνατόν περισσότερου από εσά στο σεμινάριο που θα λάβει η χώρα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σα και προσβλέπω στις ερωτήσει σα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ για όλα αυτά που μας ε, είπατε. Και επίσης και για το ότι μας συγχαρήκατε για την εκλογή μας. Ε, τώρα μπορεί να ξεκινήσει η συζήτηση. Μέχρι τώρα έξι έχουν ζητήσει το λόγο. Ε, ξεκινάει η κυρία Εκ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση που μας κάνατε σχετικά με τις προτεραιότητες της Ζωηδικής Προεδρίας. Ε, για τα δικά μου τουλάχιστον αυτιά δεν αποτελούν έκπληξη αυτά που μου είπατε, τα έχω ξανακούσει με Αλλά έχω δύο δύσκολα μεν σημαντικά δε θέματα να θίξω. Πρόσφατα εγκρίναμε μία έκθεσή μου για τον προπολογισμό και σημειώνουμε ότι το Συμβούλιο προτείνει περικοπές ε, στον ε, προπολογισμό ε, για την έρευνα. Περικοπές που κυμαίνονται από 6 μέχρι 59%. Γνωστή συζήτηση και γνωστό πρόβλημα γιατί με τις δημοσιονομικές προοπτικές που συμφωνήθηκαν για την περίοδο αυτή υπήρξε πρόβλημα το οποίο επιλύθηκε τελευταία στιγμή. Το Κοινοβούλιο προτείνει αυξήσεις, η μείωση των περικοπών, οπότε κάποια στιγμή θα πρέπει να το βρούμε. Τώρα, το άλλο θέμα είναι η γραφειοκρατία. Δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα εν μία νυχτή ή τέλος πάντων μέχρι το Δεκέμβριο. Μπορούμε όμως να, να κάνουμε κάποια βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Τον Αύγουστο ε, συμμετείχα σε κάποιες ε, διασκέψεις με τη συμμετοχή των επιχειρήσεων και διαπίστωσα ότι πολλές από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στην παγκόσμια σκηνή δεν ασχολούνται καν, δεν μπαίνουν καν στον κόπο να υποβάλουν αίτηση ε, για συμμετοχή σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Και αυτό λόγω της γραφειοκρατίας και των καθυστερήσεων που αυτή προκαλεί. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε κάτι γι' αυτό τώρα, τους επόμενους μήνες, να βελτιώσουμε την κατάσταση υπό τα δύο αυτικά, αυτά πρίσματα. Vážený pane ministře, děkuji za Ευχαριστώ πολύ. Μιλήσατε για την σημασία που έχει η δημιουργία μιας ε, συνεργασίας ε, με τη συμμετοχή όλων των αρμοδίων ε, φορέων, των πολιτών, της επιστημονικής κοινότητας και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Η συμμετοχή των κρατών μελών σε αυτό το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο και ο αριθμός των προγραμμάτων μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα λεγόμενα νέα κράτη-μέλη στα... στο 7ο πρόγραμμα, ε, πρόγραμμα πλαίσιο συμμετέχουν λιγότερο από ό,τι τα παλαιά. Υπάρχει λοιπόν μια έλλειψη ισορροπίας, μια αναντιστοιχία. Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό οι ερευνητές ε, από τις νέες χώρες ε, μετακινούνται λιγότερο, ε, δεν ξέρω. Ίσως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο δρόμο που οδηγούν στη συμμετοχή, στο που οδηγεί στη συμμετοχή στα προγράμματα αυτά να είναι μεγαλύτερα. Ίσως αυτά τα εμπόδια να οφείλονται ε, και στη δική μας ε, γραφειοκρατία η διαδικασία. Είπε λοιπόν η Σουηδική Προεδρία ότι κάποια από αυτά τα εμπόδια θα πρέπει να αρθούν, κάποιοι από αυτούς τους φραγμούς θα πρέπει να πέσουν, ούτως ώστε η συμμετοχή στα ερευνητικά προγράμματα να είναι μεγαλύτερη. Ναι, αλλά πώς. Eh, eh, Καλημέρα κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι η πρώτη φορά ως νεοεκλογήσα, νεοεκλεγήσα βουλευτής που λαμβάνω το λόγο. Δράτω με τις ευκαιρίες για να σας χαιρετήσω όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τον κύριο Υπουργό για την παρουσίασή του και να κάνω ένα σχόλιο και μία ερώτηση. Sobre Πάντα για την καινοτομία. Στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης που διάγουμε, αλλά και της προσπάθειας καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών, σε σχέση με την ε, έρευνα και τεχνολογία θα πρέπει να έχουμε μια οικονομικά βιώσιμη ε, ε, προσέγγιση. Η καινοτομία, η καινοτομία είναι μια δραστηριότητα που θα πρέπει να θέσουμε να φέρουμε σε πέρας, ιδιαίτερα για να επιλύσουμε τα προβλήματα των ε, ε, ενεργοβόρων επιχειρήσεων και μορφών κατανάλωσης. Γι' αυτό εξάλλου υπάρχει αυτό το πακέτο καινοτομία. Η ερώτησή μου. Ποια είναι τα σχέδια της ε, Προεδρίας για να δώσει νέα όθηση σε αυτό το πακέτο και να υποστηρίξει όλες τις δράσεις ε, καινοτομίας. Και στην καινοτομία όχι μόνο που βασίζεται στην έρευνα, αλλά μια γενικότερη καινοτομία, νέες μορφές καινοτομίας. Κοινωνική καινοτομία, καινοτομία στην παρέμβαση του δημόσιου τομέα, θα ήθελα λοιπόν κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες ό,τι αφορά την καινοτομία γενικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κυρία Ριέρα Μαντουρέρα. Eh, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε. Του ευχαριστώ πολύ τον εκπρόσωπο της Σουηδική Προεδρίας για την παρουσία του εδώ, αλλά και την παρουσίαση που μα έκανε των προτεραιοτήτων της Σουηδική Προεδρίας για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως η έρευνα που αποτελεί ένα από τα δυνατότερα όπλα που έχουμε στη διάθεσή μας για να εξέλθουμε της κρίσεως. Η έρευνα με, μαζί με την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία ήταν πάντα σημαντικά όπλα Το είπε και ο Υπουργό. Ε, σήμερα το είπαμε και εμεί στην πρωινή συζήτηση που είχαμε για τον προπολογισμό. Αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι στην πράξη η καινοτομία ε, έχει λιγότερη σημασία στην ατζέντα των πολιτικών ηθινόντων, αλλά και υπό όρου προπολογισμού. Τι μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε το όλο αυτό πλαίσιο. Είπατε για μεγαλύτερο συντονισμό, είπατε ε, αναφέρεται το τρίγωνο της γνώσης, ε, τα ποιότητα των πανεπιστημίων. Σωστά, σωστά. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να ασχοληθούμε στην πράξη με το θέμα αυτό και όχι μόνο θεωρητικά. Να δούμε δηλαδή τι πρακτικά βήματα μπορούμε να κάνουμε εάν θέλουμε πραγματικά όπως έλεγε η συναδελφός μου χτες, Αντριάν Αντικάου, εάν πραγματικά θέλουμε, λέγω, η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελέσει μια οικονομία που να βασίζεται στην γνώση, να είναι δυναμική τε και ανταγωνιστική. Τούτων λεχθέντων, ε, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας υποβάλω δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πρώτη, για τον ε, κανονισμό που αφορά τις υποδομές για την ευρωπαϊκή έρευνα που εγκρίθηκε από αυτήν την ε, Επιτροπή στην προηγούμενη θητεία και για την οποία ήμουν εισηγήτρια. Το Κοινοβούλιο, κύριε Υπουργέ, έκανε τη δουλειά του, νομίζω καλά, με την ε, συνεργασία όλων των ε, πολιτικών ομάδων. Μια διαβούλευση ήταν ουσιαστικά αυτή η δουλειά, διότι μόνο συμβουλευτικό ρόλο είχαμε, ζητήσαμε πιο σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουμε, αλλά δεχτήκαμε αυτόν τον συμβουλευτικό ρόλο λόγω των δεσμεύσεων που είχαμε εκ των προτέρων ε, αναλάβει. Και αργότερα μάθαμε ότι δεν εγκρίθηκε το θέμα λόγω προβλημάτων στο Συμβούλιο, προβλημάτων ΦΠΑ ελήθησαν αυτά τα προβλήματα και αυτό το καλοκαίρι, κατά τη διάρκεια της δικής σας λίγη δηλαδή Προεδρίας, ξεκίνησε. Αυτό το Κοινοβούλιο και αυτή η Επιτροπή μέχρι τώρα όμως δεν έχει καμία πληροφορία επί του θέματος. Αγνοούμε πώς επιλύθηκε τελικά ο κόμβος αυτός, το πρόβλημα αυτό και πώς ξεκίνησε να εφαρμόζεται σε ορισμένες συγκεκριμένες ε, περιπτώσεις όπως ας πούμε το πρόγραμμα που θα εγκατασταθεί στη χώρα σας και αφορά τα νετρόνια. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω την άποψή σας αν αυτή η μορφή που επιλέξατε, δηλαδή μέσω του άρθρου 161, είναι η πλέον χρήσιμη. Και ένα δεύτερο ερώτημα. Αναφέρατε στην παρουσίασή σας δύο θέματα, δύο φακέλους που θα μας απασχολήσουν και μας. Το Alzheimer και άλλες ε, ε, νευρολογικές ασθένειες. Γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το joint programming και όχι τον κοινό προγραμματισμό, δηλαδή και όχι κατευθείαν το άρθρο 169. Η ερώτησή μου είναι πώς αξιολογείται αυτό το νέο μέσο, τον κοινό προγραμματισμό, το joint programming. Και να σας πω επίσης ότι εμείς, η Επιτροπή δηλαδή αυτή, για τα δύο αυτά θέματα θα προτιμούσαμε να περάσουν από το άρθρο 169 για να μπορέσει έτσι το Κοινοβούλιο να έχει σημαντικότερο λέγειν για τα τόσο σημαντικά αυτά θέματα. Και τέλος, θα ήθελα να σας ζητήσω περισσότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα της πρόσφατης διάσκεψης που έλαβε χώρα στο Γκέτεμποργκ για το τρίγωνο της γνώσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία συνάδελφε. Γιώργο Σίσιλη και μετά θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα πριν ε, μια μικρή διακοπή για να απαντήσει ο Υπουργός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα αυτή παρουσίαση. Το ερώτημά μου αφορά το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Έχουμε αποκτήσει περισσότερη εμπειρία και με ενημερώνουν τώρα ερευνητές πως είναι ακόμη δυσκολότερο να αντλήσει κανείς κονδύλια γιατί υπάρχει ακόμη μεγαλύτερο διοικητικό βάρος. Θυμάμαι πως ε, ε, μία από τις βασικές απαιτήσει ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά ήταν να μειωθεί το διοικητικό βάρος. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω τι θα κάνει η Σουηδική Προεδρία έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται πιο αποτελεσματικά τα ερευνητικά κονδύλια, να μειωθεί επιτέλους πραγματικά η γραφειοκρατία. Τι σκοπεύετε να κάνετε έτσι ώστε να είναι πιο προσβάσιμα και για μικρότερες ερευνητικέ ομάδες τα κονδύλια. Δεύτερον, αναφέρατε το τρίγωνο της ε, γνώσης πολλές φορές ε, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας συστάθηκε και ένα τεχνολογικό Ινστιτούτο. Θα ήθελα να γνωρίζω τι πρόοδο αναμένει η Σουηδική Προεδρία στον τομέα αυτόν. Τρίτο ερώτημα. Πού βρίσκεται στον κατάλογο προτεραιοτήτων σας η έρευνα όταν σκεφτόμαστε και σκέφτεστε και εσείς τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να δώσω την ευκαιρία στον κύριο Υπουργό να απαντήσει. Ήταν σύντομε οι ερωτήσεις οπότε έχουμε και ε, λίγο χρόνο. Κύριε Υπουργέ, λοιπόν, έχετε τον λόγο να απαντήσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πραγματικά απόλαυση να βρίσκομαι στην Επιτροπή σας, καθώς είστε και πολύ παθιασμένοι για αυτό τον τομέα και υπάρχουν πολλά συναρπαστικά ζητήματα που θα μας απασχολήσουν. Ελπίζω λοιπόν να δώσω όσο δυνατόν περισσότερες απαντήσεις. Κοιτάξτε, εγώ είμαι Ερευνητή είμαι ο ίδιος πανεπιστημιακό, οπότε είναι και για μένα σημαντικό να μειωθεί η γραφειοκρατία, να γίνουν τα πράγματα πιο απλά για την έρευνα. Οπότε λαμβάνομαι τις απόψεις που ακούστηκαν. Εμείς ε, επιφέραμε κάποιες μεταρρυθμίσεις ε, για να γίνει πιο εύκολο να ζητήσουν οι ερευνητέ κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζω να συνεχιστούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις. το θέμα του προϋπολογισμού τώρα. Όπως σας είπα στην αρχική μου δήλωση, η Σουηδοί είναι διάσημη για το ότι θεωρούν ότι πρέπει να δίνουμε πολλά χρήματα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ε, έρευνα, π.χ. μπορούν να φύγουν κονδύλια από τη Γεωργία. Αυτή είναι η θέση μας, αλλά πρέπει να δούμε και το τι υπάρχει αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από κονδύλια πρέπει να φροντίσουμε να βελτιώσουμε την ανάπτυξη και την έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρχει μεγαλύτερη όθηση γενικότερα να θεωρήσουμε αυτούς εταίρους στην ερευνητική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε λοιπόν φιλοδοξίες και θέλουμε να κάνουμε μια διαφορά στο μέτωπο αυτό κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Όσον αφορά τώρα την ε, διανομή των κονδυλίων από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό Έρευνας και το πώς διανέμονται αυτά στα διάφορα κράτη-μέλη. Νομίζω πως είναι σημαντικό εδώ να σημειώσουμε πως ε, Πρέπει να δουλέψουμε με τους κανονισμούς ε, που έχουμε, θα ισχύσουν για πολλά χρόνια ακόμα, αλλά η Κομισιόν βεβαίως μπορεί να επιφέρει κάποιες αλλαγές εάν ε, είναι αυτό απαραίτητο. Έχουμε ένα σύστημα, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε μέχρι να λάβουμε απόφαση για το μελλοντικό σύστημα. Οπότε οι κανόνες είναι αυτοί που είναι. Το τρίγωνο της γνώσης τώρα που ανέφεραν αρκετοί. προσπαθούμε εμείς με αυτόν τον τρόπο να περιγράψουμε πόσο σημαντικό είναι να σημειωθεί πρόοδο στην πολιτική καινοτομία. Είχαμε μια σημαντική διάσκεψη και χαίρομαι που θα προσπαθήσουμε με ενθουσιασμό να προωθήσω αυτά τα ζητήματα τους ερχόμενου μήνες. Τώρα ήταν και κάτι που το είχαμε υποσχεθεί. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες που πρέπει να εκμεταλλευτούμε και θεωρούμε πως ο κοινός προγραμματισμός είναι κλειδί στον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας και για να αναπτυχθεί αυτός ο χώρος θεωρούμε πως η συνεισφορά και η βελτίωση της έρευνας στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντική ειδικά αυτή τη στιγμή κατόπιν όσον αφορά τις ε, πληροφορίες που δίδονται στο Κοινοβούλιο συγκεκριμένα κατά περίπτωση. Οπωσδήποτε θα ερχόμαστε από το Συμβούλιο να σας ενημερώνουμε. Σας ευχαριστώ. Αρχίζει η επόμενη ομάδα. Νίμπλερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, χαίρομαι που ήρθατε στην Επιτροπή μας ε, και θα έχετε μαζί μας ε, το διάλογο για την πολιτική έρευνα και για τα βασικά θέματα της Προεδρίας σας. Υπάρχουν δύο θέματα που θέλω να θίξω. Βεβαίως, εν μέρη έχω ήδη καλυφθεί η πολιτική έρευνα στα τελευταία χρόνια, εγώ στο Κοινοβούλιο είμαι εδώ και 10 χρόνια, καταλαμβάνει όλο και μεγαλύτερη σημασία. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια προετοιμασία των απαραίτητων δομών και είπατε κι εσείς ε, ότι αυτή τη στιγμή τρέχουν κοινά προγράμματα. Αυτά τα βρίσκω πολύ καλά. Το γεγονός ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνεργαζόμαστε περισσότερο και με τον τρόπο αυτό αποφεύγουμε και επικαλύψεις στα μεμονωμένα κράτη-μέλη. Στις συζητήσεις που είχαμε με τους ε, συναδέλφους μου, ε, συναδέλφους από το Bundestag της Γερμανίας, ακούω πάρα πολλές επιφυλάξεις, γιατί πολλοί φοβούνται ότι εδώ παρεμβαίνουμε σε θέματα εθνικής ε, κυριαρχίας. Και θέλω να ρωτήσω το εξή. Εσείς ε, έχετε συζητήσεις με τα 26 κράτη-μέλη και ρωτώ, και εσείς έχετε συναντήσει επιφυλάξεις, έχετε διαπιστώσει ότι υπάρχουν εμπόδια έτσι ώστε να υπάρξουν κοινοί οργανισμοί, κοινά προγράμματα και κοινέ υποδομές στην έρευνα. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Και η δεύτερη αφορά στο ε, ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο. Είπατε σωστά ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι προετοιμασίες Πώς θα μοιάζει λοιπόν το 8ο. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 7ο. Να μην πω ότι έχουμε και το 6ο που και αυτό ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Ερωτώ λοιπόν, από πλευρά των κρατών μελών υπάρχουν κάποιες σκέψεις για το πού θα δοθεί το βάρος στο 8ο πρόγραμμα πλαίσιο. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τις συζητήσεις που είχαμε εδώ κατά την έγκριση του 7ου προγράμματος ε, πλαίσιο. Είχαμε πει να περιοριστεί η γραφειοκρατία, να διευκολυνθούν οι μειοδοτικοί διαγωνισμοί και με ενδιαφέρει να μας πείτε ποιες είναι οι συγκεκριμένες προτάσεις. Και εδώ αναφέρομαι και στον πρόεδρο της Επιτροπής μας. Ίσως του χρόνου θα μπορούσαμε να προσκαλέσουμε ερευνητές στην Επιτροπή μας, οι οποίοι ακριβώς θα μας αναφέρουν τι ακριβώς έχει βελτιωθεί με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Γιατί πριν από λίγα χρόνια ξεκινήσαμε φιλόδοξα, θέλαμε να περιορίσουμε την γραφειοκρατία, να πλουστεύσουμε τις διαδικασίες και εγώ Ρωτώ λοιπόν και πάλι ε, στο 8ο πρόγραμμα πλαίσιο που θα δώσετε βάρος. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο πρόεδρος, ο συνάδελφος Ρούντι. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσία σας εδώ και τις ε, πληροφορίες και τις πολιτικές ενδείξεις που μας δώσατε. Δύο ε, ερωτήσεις και ένα σχόλιο. Η ερώτηση. Είπατε προηγουμένως ότι θα πρέπει να έχουμε μια μακροπρόθεσμη θεώρηση των πραγμάτων. Σωστό. Διότι οι πολίτες ε, αυτό περιμένουν από εμά Να δώσουμε θετική όθηση στις ε, εξελίξεις του μέλλοντος. Και για το κράτος μέλος το οποίο ανήκετε, αλλά και ως ασκόν την ε, Προεδρία. Πιστεύετε ότι η έρευνα μπορεί να είναι ο τομέας ο που όπως κάναμε με την κοινή αγροτική πολιτική μπορούμε να ομογενοποιήσουμε τα κονδύλια δεν θα μπορούσε να γίνει η νέα πραγματικά μεγάλη κοινή πολιτική της Ένωσης. Πολιτικά δεν θεωρείτε ότι αυτή η ιδέα είναι καινοτόμος. Το σχόλιο Νομίζω ότι κοινό σημείο σε όλες τις των Σανδέρφων είναι η γραφειοκρατία της ε, λειτουργίας της Ευρώπης, εις ό,τι αφορά την διανομή, την έγκριση και τον επιμερισμό των κοντιλίων στα ερευνητικά κέντρα. Ε, ψηφίσαμε μια τροπολογία της κυρίας Κράσλο για να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να άρει μια σειρά εμποδίων ε, γραφειοκρατικής ε, φύσεως, εσωτερικών ελέγχων ε, που αποτελούν επικάλυψη τα μεν με τα δε κάτι το οποίο κάνει τους ερευνητές να απαυδίσουν, να σηκώσουν τα χέρια ψηλά και τελικά να αδιαφορήσουν μακροπρόθεσμα για τις δυνατότητες που δίνει η Ένωση. Εφιστώ την προσοχή σας επ' αυτό, διότι θα θέλαμε συλλογικά, όχι μόνο εμείς ως Επιτροπή, όχι μόνο ως Κοινοβούλιο, συλλογικά όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να ζητήσουν από την ε, Κομισιόν να διευκολύνει τη διαδικασία προς χάρη των επιχειρήσεων, ε, κάτι εξάλλου που είναι και το ζητούμενο. Ευχαριστώ. Colegin Ticău. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Conform strategiei de la Lisabona, statele membre ar trebui... Σύμφωνα με τη στρατηγική της Λισαβόνας, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αφιερώσουν στην έρευνα το 3% του ΑΕΠ τους. Αυτό το, από αυτό το ποσό, τα δύο τρίτα, πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα. Το ερώτημά μου, δεδομένου ότι η έρευνα και η ανάπτυξη αφασίζονται στην παιδεία, το ερώτημά μου, λοιπόν, ποια μέτρα δεδομένης και της οικονομικής κρίσης ε, στην οποία βρισκόμαστε ποια μέτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν δεδομένης και της μείωσης ε, του ΑΕΠ των κρατών μελών λόγω της κρίσης. Ποια είναι λοιπόν τα μέτρα που προβλέπετε για να αναζωογονήσετε τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και ε, να αυξήσετε τις επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και κυρίως της εφηρμοσμένης έρευνας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Μιλώ υποδιπλή ιδιότητα και ως Ευρωβουλευτής αλλά και ως πανεπιστημιακός. Το πανεπιστήμιό μου έχει συμμετάσχει σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα και γι' αυτό θα ήθελα να μιλήσω αυτή τη, υπό αυτή την διπλή ιδιότητα. Γνωρίζω λοιπόν τα των πανεπιστημίων και της έρευνας και πιστεύω ότι αλλάζουν υπερβολικά τα πράγματα όταν αλλάζει το κάθε πρόγραμμα πλαίσιο. Στο πέμπτο πρόγραμμα πλαίσιο δίδαμε έμφαση στα μικρά προγράμματα. Στο έκτο ισορροπήθηκαν τα πράγματα μεταξύ μικρότερων και μεγαλύτερων δικτύων. Στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο δώσαμε έμφαση στα μεγάλα προγράμματα και στη δικτύωση και οι ερευνητές ε, κάποια στιγμή σηκώνουν τα χέρια ψηλά διότι ε, δεν μπορούν να έχουν μια συνέχεια στο έργο τους. Είναι επίγον λοιπόν όταν αναδιατυπωθεί το νέο πρόγραμμα πλαίσιο να καθορίσουμε άπαξ και διαπαντός ποια είναι τα μέσα που έχουν στη θέση τους οι επιστήμονες, οι ερευνητές διότι όταν αλλάζουν τα πράγματα κάθε τρεις και λίγο αυτό μόνο κακό κάνει. Τώρα, με κάθε αλλαγή πρέπει να, μαθαίνουμε, να μαθαίνει κανείς εκ νέου πώς θα χρησιμοποιήσει τη διαδικασία. Από το μηδέν. Φτού και από την αρχή δηλαδή. Αυτό θεωρώ ότι αποτελεί μια πολύ μεγάλη δυσκολία που ε, αντιμετωπίζουν ε, οι ερευνητές. Και έχει να κάνει και με τη γραφειοκρατία, διότι περί γραφειοκρατίας πρόκειται είναι προγράμματα όπως το Science Society ας πούμε το οποίο αλλάζει υπερβολικά συχνά τις απαιτήσει του, τις προδιαγραφές του, το περιεχόμενό του γιατί δεν μπορούμε, αυτό δεν μπορούμε λοιπόν να το δεχθούμε. Δεν μπορούμε να δείχνουμε τέτοια έλλειψη συνέπειας. Δύο ερωτήματα ή δύο θέματα αν θέλετε. Οι προτεραιότητες στον τομέα της έρευνας. Ο... Μιλήσατε κύριε Υπουργέ για την προτεραιότητα που αφορά την ασθένεια του Αλτσχάιμερ και άλλων νευρολογικών ασθενειών. Είχαμε άλλες προτεραιότητες, νανοτεχνολογία, γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί κτλ. Για τις ερευνητικές ομάδες, για τα δίκτυα, οι προτεραιότητες ε, θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο συνένεσης μεταξύ όλων των ε, εμπλεκομένων φορέων. Προφανώς και κατανοώ και δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό ότι οι προτεραιότητες αυτές ε, είναι καρπός μιας πολιτικής προσέγγισης, αλλά μόνο όταν είναι συνενετικοί αυτοί οι στόχοι θα μπορέσουν οι επιστήμονες να τα βγάλουν πέρα και αφορά κάθε πρόγραμμα και κάθε κύκλο στον οποίο εντάσσονται τα προγράμματα. Ένα ακόμα σχόλιο για τις τρίτες χώρες. Υπάρχουν διάφορα εργαλεία και μέσα που μας δίδουν την δυνατότητα να, να δώσουν δυνατότητα σε ερευνητές από τρίτες χώρες να συμμετάσχουν ε, στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Βεβαίω η γραφειοκρατία είναι ακόμα μεγαλύτερη, αλλά δεν ήθελα να σχολιάσω αυτό. Ήθελα να σχολιάσω το εξή. Πρέπει να ενδυναμώσουμε, να ενισχύσουμε τον ευρωπαϊκό ερευνητικό χώρο. Πώς γίνεται αυτό, με ομφαλοσκόπηση ή με άνοιγμα προς τα έξω, με άνοιγμα προς τον κόσμο. και εδώ δεν ακολουθούμε μια συνεπή στάση. Άλλες φορές είμαστε κλειστοί, σε άλλους τομείς ομφαλοσκοπούμε, σε άλλους τομείς ε, ανοιγόμαστε περισσότερο. Δεν θα πρέπει λοιπόν, αυτή είναι η ερώτησή μου, να επιλέξουμε μία στάση. Έχω πολλά ακόμα να πω, θα είχα πολλά ακόμα να πω, θα είχα Πολλέ ερωτήσει να θέσω για την πρακτική εφαρμογή του 7ου προγράμματος πλαισίου, γι' αυτό σταματώ εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Στάλφος ε, Λάμπαρτς. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, πρώτα απ' όλα, ως ε, πράσινος ε, θέλω να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που αναφερθήκατε στις ε, προτεραιότητες της Ιουδικής Προεδρίας που ταιριάζουν πάρα πολύ καλά με το δικό μας το πρόγραμμα και που ε, χρειάζεται πραγματικά αυτό που αναφέρετε για να αντιμετωπίσουμε και τις οικονομικές αλλά και τις κλιματικές ε, προκλήσεις. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μόνο το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, εξαντλούνται και οι πόροι. Επειδή λοιπόν είμαστε εδώ ένα μικρό ακροατήριο, θα ήθελα να έχω την άποψή σας ε, ως Υπουργού αλλά και ως Ακαδημαϊκού για τρία θέματα. Πρώτον, αναφερθήκατε στην αποτελεσματικότητα αυτών που καταναλώνουμε. Και είναι αλήθεια ότι αν θέλουμε να δαπανίσουμε περισσότερα για την έρευνα, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι γίνεται και σωστή χρήση των κονδυλίων. 100% αποτελεσματικότητα, αυτό είναι ουτοπικό, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν μπορούσατε κάτι να κάνατε, πού θα ξεκινάγατε για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα στην έρευνα. Δεύτερον, την ίδια ερώτηση θέλω να κάνω για την πρόσβαση των ΜΜΕ. Ε, εκεί παίζει ρόλο η καινοτομία. Κάποιοι λένε ότι χρειαζόμαστε την ε, κρίσιμη μάζα ε, και ότι οι αλλαγέ μπορούν να γίνουν μόνο σε μεγάλου φορεί. Άλλοι πάλι λένε ότι οι καινοτόμε ιδέε μπορούν να ανθίσουν μόνο σε μικρέ επιχειρήσει. Ποια είναι η δική σα άποψη από αυτού. Οι μικρομεσαίες έχουν πρόβλημα στο να έχουν πρόσβαση στα κονδύλια. Αναφέρομαι σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, αλλά και σε μικρά εργαστήρια ενδεχομένω, που και αυτά μπορεί να έχουν πρόβλημα απόκτησης κονδυλίων. Εσείς τι πιστεύετε, ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ε, θέλουν να προβούν ε, σε καινοτομίες ε, και αν ναι, τότε πώς γίνεται αυτό. Και τελευταία μου ερώτηση. Θα ήθελα πάλι την προσωπική σας άποψη για το εξής. Αυτό από το οποίο υποφέρουμε στην Ευρώπη είναι η διασπορά, η διάχυση των προσπαθειών μας. Διαχέονται οι προσπάθειες σε διάφορες προτεραιότητες και ούμον αυτό, αλλά και σε διάφορες χώρες, 27. Ε, δύσκολο λοιπόν να επιτύχει κανείς την κρίσιμη μάζα. Ε, κατά τη δική μου άποψη, τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μπορούν να είναι καταλυτικά. Δεν είναι ο μόνος τρόπος, μπορούν όμως να αποτελέσουν ένα είδος καταλύτη. Και κατά την άποψή σας, πώς μπορούμε να επιτύχουμε βελτίωση. Και άλλο ένα τελευταίο σχόλιο. Εσείς είσαστε αρμόδιους για την έρευνα και έχετε τους συναδέλφους σας, υπουργούς έρευνας. Πώς πιστεύετε ότι μπορούμε εμείς να μετρήσουμε στους συναδέλφους μας για να μας αναγνωρίζουν περισσότερο. Ποιο είναι το βάρος μας. Πιστεύετε ότι οι συνάδελφοί σας σε άλλα υπουργεία την έρευνα την αντιμετωπίζουν ως ένα στρατηγικό κεφάλαιο για να βρούμε μια διέξοδο από την κρίση ο επόμενος ε, συνάδελφος και ζητώ συγγνώμη αν η προφορά μου δεν είναι και σωστή. Ε, Αξιότιμε Υπουργέ, θα ήθελα ευθύ εξ αρχή ε, να σα ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας σήμερα στην Επιτροπή. Μιλάμε για τα ερευνητικά προγράμματα. Τόσο εμείς όσο και τα κράτη-μέλη ξέρουμε βέβαια πολύ καλά ότι υπάρχει ένας φαύλος κύκλος. Λόγω της ε, κρίσης, της χρηματοπιστωτικής, είναι δύσκολο να λύσουμε και το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και της κατανάλωσης ενέργειας. Η επίλυση των ενεργειακών προβλημάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις ε, νυν και μελλοντικές επενδύσεις. Το κόστος θα είναι υψηλό, αλλά απαιτείται και στενή συνεργασία στον τομέα της ε, έρευνας. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα στα 27 κράτη-μέλη. Και τα περισσότερα από αυτά τα προβλήματα εμφανίζονται στα αποκαλούμενα νέα κράτη. Τα προβλήματα αυτά ανάγονται στο παρελθόν αυτών των κρατών και σήμερα χαίρομαι που είμαι στην ευχάριστη θέση που χαίρομαι που από αυτά που μας είπατε, ορισμένες χώρες, κυρίως οι χώρες της Βαλτικής, ε, αντιμετωπίζονται πολύ θετικά από εσάς. Είπατε ότι η Βαλτική θα είναι προτεραιότητα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Μήπως μπορείτε λιγάκι να το συγκεκριμενοποιήσετε αυτό. Αναφέρομαι πάντα στις χώρες της Βαλτικής. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ε, Γκρίφτον. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Λάμπερτ για τους πόρους. Θα γνωρίζουν πολλά μέλη της ε, Επιτροπής πως ε, πολλές από τις νέες ε, τεχνολογίες στις οποίες βασίζουμε τις ελπίδες μας βασίζονται σε σπάνια στοιχεία όπως το λίθο παραδείγματος χάρη που έχουν αστρονομικές τιμές. Αυτό το οποίο όμως δεν είναι γνωστό είναι ότι 95% των σπανίων μετάλλων του κόσμου παράγονται στην Κίνα και η Κίνα σχεδιάζει να περιορίσει ή και να απαγορεύσει την εξαγωγή τους. Οπότε θα μειωθεί η δυνατότητα να κάνουμε εμείς έρευνα σε αυτό το ζωτικό τομέα. Μπορεί ο κύριος Υπουργός να μας πει τι σκοπεύει να κάνει για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα και συγκεκριμένα εάν η, Κιν, η Προεδρία με συγχωρείτε σκοπεύει να διεξαγάγει ένα διεθνή έλεγχο για την ύπαρξη των σπανίων μετάλλων αλλά και των αποθεμάτων πετρελαίου έτσι ώστε οι αποφάσεις μας ε, να βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία για να ξέρουμε πότε θα φτάσουμε στην κορύφωση της παραγωγής πετρελαίου εάν δεν την έχουμε ήδη φτάσει και αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτή η τρομακτική έλλειψη πρώτων υλών για τον βιομηχανικό μας ε, πολιτισμό. Σας ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Υπουργό. Για το πρόβλημα της ε, έρευνας θα ήθελα να θίξω ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι δεν αναφέρθηκε από τους λοιπούς συναδελφούς. Εσείς ευχηθήκατε, αναφέρατε ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συνένεση, μεγαλύτερη συμμετοχή στη συνενετική διαδικασία όλων των εμπλοκομένων φορέων. Όπω το Κοινοβούλιο, που δεν συμμετείχε πάντα στι διαβουλεύσει για το καθορισμό του προηγούμενου του προγράμματο γιατί είπατε ότι οι προτεραιότητες έτσι θα είναι πιο συνεννοητικές, όλοι θα συμφωνούν για την επιλογή αυτών των προτεραιοτήτων. Πιστεύω ότι είναι απόλυτα σωστή αυτή η άποψη, αυτή η καινοτόμος, γιατί περί αυτού πρόκειται προσέγγιση Πώς θα το επιτύχετε αυτό. Οποιαδήποτε σας ε, πρόταση προς αυτήν την κατεύθυνση προφανώς εμάς μας βρίσκει συμφώνους. Ευχαριστώ. Αυτή ήταν η τελευταία τοποθέτηση οπότε τώρα ο κύριος Υπουργό έχει την ευκαιρία να απαντήσει σε αυτές τις ωραίες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω πως ε, θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα βασικά ζητήματα που ανέφεραν οι προλαλήσαντες. Κοιτάξτε, υπάρχει εδώ πέρα μια δύσκολη ισορροπία μεταξύ της ευρωπαϊκής πολιτικής ε, έρευνας και των επενδύσεων που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και των επενδύσεων που γίνονται σε επίπεδο κράτους μέλους. Πρέπει να βρούμε λοιπόν μια ισορροπία να διορθεί αυτό το πρόβλημα και αυτό θα γίνει με τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Πρέπει να συνεργαστούμε λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με τα κράτη-μέλη χωρίς να υποθέτουμε πως ε, θα περάσουν όλες οι εξουσίες στην Κομισιόν ε, στις Βρυξέλλες γενικώ όπως κάποιοι νομίζουν. Αλλά νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βρούμε την ισορροπία την ευαίσθητη μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κράτους μέλου όσον αφορά τις επενδύσεις. Όσον αφορά το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο, εμείς θέλουμε να ξεκινήσει η συζήτηση κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Προφανώς θα συνεχίσει και μετά από αυτήν, αλλά θέλουμε να συζητήσουμε τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη και στον κόσμο, όπως η κλιματική αλλαγή, παραδείγματο χάρη. Οι σοβαρές ασθένειε πανδημίες, ε, και τα λοιπά. Ως ανθρωπότητα συνολικά αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα και τέλος κάποιος ανέφερε και τη χρηματοδότηση. Και εδώ, όπως ανέφερα, νομίζω ότι συμβαίνει το εξής. Στην Σουηδία έχουμε σαφή θέση. Ο Ευρωπαϊκός υπολογισμό έρευνα μακροπρόθεσμα πρέπει να αυξηθεί. Τα χρήματα πρέπει, εμείς λέμε, να έρθουν από τη γεωργική πολιτική και σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να συντονίσουμε τους πόρους που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και πάλι, όπως σας είπα, ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας είναι ο τρόπος για να το επιτύχουμε αυτό. Όπως σας είπα, είμαι πολύ ικανοποιημένο από τα σχόλια που ακούστηκαν για τη γραφειοκρατία. Όπως σας είπα και εγώ είμαι ερευνητής ε, και ακόμα και στο εθνικό επίπεδο είχα προβλήματα με τη γραφειοκρατία και αντιλαμβάνομαι πως στην Επιτροπή εδώ πέρα μιλάμε για την ευρωπαϊκή γραφειοκρατία που αντιμετωπίζει η έρευνα αλλά υπάρχει αυτό το πρόβλημα σε όλες τις ε, χώρες μας και οπωσδήποτε στη Σουηδία το έχουμε αυτό το πρόβλημα και πρέπει να προσπαθήσουμε να το επιλύσουμε και διαπιστώνω πως έχετε σαφή δέσμευση για αυτό το θέμα είναι προτεραιότητα της Σουηδικής Προεδρία θέλουμε να περάσουν τα πράγματα. Θέλουμε να περάσουν κάποια πράγματα από αυτή την Επιτροπή για να βελτιωθεί η κατάσταση της γραφειοκρατίας, γιατί θα υπάρξει κάποια αντίσταση, οπότε αναμένω να με βοηθήσετε σε αυτή τη μάχη όσον αφορά τον στόχο του 3% για επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη. Είναι πολύ σημαντικός. Έχουν γίνει κάποιες αξιολογήσεις. Δεν έχουμε προχωρήσει τόσο όσο θα θέλαμε πρέπει να διασφαλίσουμε πως ε, θα αυξηθεί ο ρυθμός για να φτάσουμε το 3%. Πολλά νέα κράτη-μέλη έλαβαν ε, σημαντικά μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση και βλέπω πως πολλές χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη επενδύουν τώρα στην έρευνα και την ανάπτυξη και ελπίζω πως θα μπορέσουμε να φτάσουμε τον στόχο του 3% και είναι σημαντικό εδώ πέρα να συνεισφέρουν και οι ιδιωτικές εταιρείε, γιατί δύο τρίτα αυτών των επενδύσεων θα έρθουν από τον ιδιωτικό τομέα και υποτίθεται πως θα είναι ε, ένα τρίτο της χρηματοδότησης, η δημόσια χρηματοδότηση. Το ερώτημα για τα διάφορα προγράμματα πλαίσιο και πώς συνδυάζονται και πώς είναι διαφορετικές προτεραιότητες είναι σημαντικό γιατί μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα για τους ερευνητές εάν δεν υπάρχει συνέχεια. και νομίζω πως ε, η βάση μιας λογικής εθνικής ή ευρωπαϊκής πολιτικής έρευνας είναι οι μακροπρόθεσμες ε, προοπτικές. Πολλές ε, μεγάλες ανακαλύψεις, καινοτομίε που ζούμε σήμερα είναι καινοτομίε που οφείλονται σε έρευνα που έγινε πριν από 30-40 χρόνια. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε μακροπρόθεσμες προοπτικές αλλά βεβαίως πρέπει να αλλάζουν και οι προτεραιότητες ε, ανάλογα με το πώς κυλούν τα πράγματα, αλλά πρέπει να το δούμε κάπως πιο μακροπρόθεσμα το θέμα της ε, ερευνητικής πολιτικής και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να επανεξετάσουμε όλα αυτά τα διαφορετικά μέσα που υπάρχουν οπότε ελπίζουμε να μπορέσουμε μακροπρόθεσμα να βελτιώσουμε την ε, νοοτροπία σε αυτόν τον τομέα. Τώρα, είναι σημαντική η... ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε όλους τους πόρους που έχουμε στην διάθεσή μας, αλλά και για να γίνουμε ενεργοί σε διεθνές επίπεδο. Οπότε αυτό αφορά την ενίσχυση του ρόλου μας και εσωτερικά, αλλά και σχέση με το τι κάνουμε με τον ε, υπόλοιπο κόσμο. Αυτό θα το επιτύχουμε με εντονότερο συντονισμό εντός της ε, Ευρώπης. Η πολιτική λοιπόν της έρευνας και η σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο αναφέρατε και ελπίζουμε πως η Κομισιόν ε, θα φέρει εδώ πέρα μια έκθεση, θα μας δώσει κάποια έμπνευση για το μελλοντικό μας έργο και τις μελλοντικέ προεδρίες γιατί δεν ξέρουμε πόσο θα προχωρήσουμε εμείς στο δικό μας εξάμεινο. Εντάξει, είμαστε φιλόδοξοι οπωσδήποτε. Κατόπιν υπάρχει και το γενικότερο ζήτημα το να πείσουμε δηλαδή τους Ευρωπαίους Υπουργούς Οικονομικών να επενδύσουν στην έρευνά και με δεδομένη την οικονομική κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε νομίζω μπορούμε να δούμε πώς γίνονται πολύ τολμηρές αποφάσεις σε κάποια κράτη-μέλη για να ενισχυθεί η έρευνα. Στη Σουηδία αυξήσαμε τις επενδύσεις κατά 5 εκατομμύρια κορώνε, δισεκατομμύρια κορώνες και πολλές ε, άλλες χώρες αυξάνουν τις προσπάθειές τους. Οπότε φαίνεται πως ε, έχουν συνειδητοποιήσει οι Υπουργοί Οικονομικών πως πρέπει τώρα λόγω της κρίσης να αυξηθούν αυτές οι επενδύσεις γιατί μακροπρόθεσμα θα ωφεληθούμε. Και βεβαίως ε, θα δούμε και τι επιρροή θα έχουν οι Υπουργοί Έρευνα στους Υπουργούς Οικονομικών. Ελπίζω να συνειδητοποιήσουν οι Υπουργοί Οικονομικών πως δεν είναι καλή ιδέα να μειωθούν παρά την κρίση οι προπολογισμοί τη έρευνα, οπότε εγώ θα καταβάλω κάθε προσπάθεια και ελπίζω να έχω και τη δική σα υποστήριξη. Τώρα, η στρατηγική τη Βαλτική και το τι γίνεται εκεί πέρα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όπω είπα στην αρχή, το πρόγραμμα Bonus είναι μια έκφραση τη προτεραιότητα που αποδίδουμε στη Βαλτική και ελπίζουμε να επιτύχουμε του στόχου σύντομα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει σύντομα και σας είμαι ευγνώμων και αναμένω και τη μελλοντική συνεργασία μαζί σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ και εξ ονόματος όλης της Επιτροπής για την επίσκεψή σας πρώτα απ' όλα, δεύτερον για τις δηλώσεις σας και τρίτον για το πόσο απατήσατε επιμελώς όλες τις ερωτήσεις. Νομίζω πως θα συνεργαστούμε καλά. Είναι εδώ πέρα ένα από τους σημαντικότερους τομείς που στους οποίους εργαζόμαστε και διακομματικά θα έλεγα γιατί μιλάμε για τους πόρους εδώ πέρα σε αυτό τον τομέα. Σας ευχαριστώ για το ότι ήσασταν τόσο σαφείς. Εύχομαι καλό ταξίδι και σας ευχαριστώ. Γεια σας. So, meine Damen Οπότε, κυρίες και κύριοι, περνάμε στο σημείο 16 διάφορα. Υποθέτω πως δεν έχετε εδώ πολλά σοβαρά πράγματα. 17 να σας πληροφορήσω πως η επόμενη συνεδρίαση είναι στις 28 Σεπτεμβρίου, 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Νομίζω χαίρεστε που θα ξανασυναντηθούμε, αλλά χαίρεστε και για το ότι τελειώσαμε σήμερα, φαντάζομαι. Εύχομαι καλή συνέχεια στι υπόλοιπε επιτροπέ ή καλό ταξίδι στο σπίτι σας. Ευχαριστώ.